Κυρίες και κύριοι, και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, Έχουν περάσει ήδη 6 λεπτά από τότε που θα έπρεπε να ξεκινήσουμε. Επομένω, α ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση αυτή. καλωσορίζω όλου στην έκτακτη αυτή συνεδρίαση Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και τη Υποπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Περνάμε στο σημείο 1, έγκριση της μερίσιας διάταξης. Υπάρχουν παρατηρήσεις. Δεν βλέπω κανέναν. Εγκρίνεται λοιπόν η μερίσια διάταξη. Περνάμε στο σημείο 2, ανακοινώσει του Προέδρου. Δεν έχω να κάνω ανακοινώσει. Επομένως μπορούμε έτσι να περάσουμε στο σημείο 3, ηλεκτρονική ψηφοφορία για την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο του 2016 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος. Η Γκοτλίβια Γκούτσπουλ Ρόβολ είναι η συγγήτρια. Θέλετε να πάρετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ξέρετε ένας πολιτικός πάντα κάτι έχει να πει κύριε Πρόεδρε. Βλέπω ότι έχουμε καλύψει τα πάντα όμως σχετικά με την έκθεση αυτή και το καλύτερο θα λοιπόν να την ψηφίσουμε τώρα. Ευχαριστούμε πολύ. Γκοντελίβε. Εγώ θα περίμενα να μιλούσε περισσότερο, γιατί περιμένω να μου φέρουν την κάρτα ψηφοφορία. Θα μου τη φέρει ο βοηθό μου. Στο ενδιάμεσο διάστημα θα έπρεπε να σας πω ότι δύο τουλάχιστον ακόμα συνάδελφοι δεν έχουν λάβει τον κατάλογο ψηφοφορία, ο κύριος Στάτνα και ο κύριος Γκάλερ. Λοιπόν, ας περάσουμε στη ψηφοφορία. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4 υπέρ. Σας ζητώ συγγνώμη, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Τροπολογία 104. Αναφέρει στη γραφή μάλιστα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 111 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 143 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 155 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Για την 155. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. 27 υπέρ, 15 κατά εγκρίνεται λοιπόν. Ο τεχνικός είναι εδώ. Ο κύριος στο βάθος έχει ένα πρόβλημα με τη συσκευή ψηφοφορίας. ...156 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Εγκρίνεται, με συγχωρείτε, διορθώνω πρόεδρος, εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται.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 Τροπολογία 229 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 230 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τροπολογία 230. Τροπολογία του κυρίου Κοράου. Άρτη ψηφοφορία. Ένα άλλος να έχει ψηφίσει ακόμα. Πολύ ωραία, πέρα. Απορρίπτεται. 18 υπέρ, 25 κατά. 231. Κόρβιν Μίκη υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 232. Σε τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, έτσι δεν είναι. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος μάλλον. Άρτη ψηφοφορία. πέρασε, Απορρίπτεται. 234 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Δεύτερο τμήμα της 234, άρτη ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. 235 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Εντάξει, ηλεκτρονική επαλήθευση για τη 235. Πρέπει να σηκώνετε και τα χέρια σας όμως, δεν σας βλέπω. Λοιπόν, άκτη ψηφοφορία τη 235. Πέρας. Εγκρίνεται. Λοιπόν, ψηφίσουμε τώρα. Συμβαστική 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 246 του κύριου Πέτ υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 259 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 21 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 282 υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 22 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 245 Σάκιο Στρεβίτσιους υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 285 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 23 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 296 του κυρίου Σαΐφ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 298 υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση για τη 298 άρθρη ψηφοφορία. Πέρας. 22 υπέρ, 21 κατά, Απορρίπτεται. «22 προς 21 είναι 22, 22 προς 23, άρα απορρίπτεται». Ψηφίσουμε τώρα τη 297 του κυρίου Πιτίδου υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 24 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 25 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 305 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η επόμενη καταπίπτει, 308 τώρα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 307 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 309 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 311 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 26 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 316 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 317 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 318 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 319 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 121 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 321 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 322 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 27 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 28 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 330 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 333 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 332 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 331 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 334 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 337 σε δύο τμήματα, λέει ο πρόεδρος. Α, συγγνώμη, συγγνώμη. 335 κοράω υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τώρα 337 υπέρ, κατά. Στο πρώτο τμήμα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Καταπίπτει το δεύτερο τμήμα γιατί εγκρίνεται 334. Τώρα. 338. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 29 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 345 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 347 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε για την 347 ηλεκτρονικά. Παρακαλώ, ψηφίστε. Πέρασε τις προφορίας εγκρίθηκε. 348 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 349 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 350 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 351 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 353 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 30 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 37. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 38 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 80 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 31 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 32 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 46 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 47 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 33 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 56 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 34 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 35 τώρα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 67 του κ. Κοράου υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 69 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 71 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την 71. Μπορείτε να ψηφίσετε. Δύο ακόμα. Άλλος ένας. Τέλος. Εγκρίθηκε. Αυτή ήταν η 71. 73 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 72 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 87 υπέρ κατά αποχές. Θα ελέγξουμε και για την 87. Παρακαλώ ψηφίστε. Ψήφισαν όλοι. Απορρίφθηκε.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 Εντάξει, ε, ό,τι θέλετε. Γκουε. Ευχαρίστω. Άλλοι τρει πρέπει να ψηφίσουν ακόμα. Ωραία, πέραση της προφορίας. 37 κατά, 8 υπέρ. Και κύριε Στέτινα, ναι, τους λάβαμε υπόψη μας. Ωραία. Λοιπόν, τώρα περνάμε στην τροπολογία 12 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 17 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 18 υπέρ,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 Αυτά. Ναι, εντάξει, μέχρι τώρα ζεσθενόμασταν. Τώρα θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά το τροποποιημένο κείμενο. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίθηκε. 41 ψήφοι υπέρ, μία ψήφος κατά. Α, 43, καλά. Η εισηγήτρια, παρακαλώ. Δύο λόγια παρακαλώ, αγαπητοί συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ θερμά για τη στήριξή σας και σας ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ γιατί τα καταφέραμε όλοι μαζί να συνεργαστούμε και να συντάξουμε μία έκθεση η οποία πραγματικά εκφράζει αυτά που θα έπρεπε να εκφράζει και επικεντρώνεται στα σημαντικά. τα καταφέραμε καλύτερα από ότι πέρυσι. Οπότε ευχαριστώ όλες τις πολιτικές ομάδες και όλα τα μέλη της Επιτροπής μας. Πρόεδρο σημείο 4, διάφορα. Παρακαλώ κύριε Ποστινάρο. Νομίζω ότι σήμερα στην ΑΦΕΤ πρέπει να μνημονεύσουμε το γεγονός ότι εγκρίθηκε η ΠΕΣΚΟ, γεννήθηκε. 23 χώρες μέλη υπέγραψαν ότι είναι έτοιμες να συμμετάσχουν στην ΠΕΣΚΟ, την Ευρωπαϊκή Άμυνα δηλαδή. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Πράγματι, ήταν μια ιστορική σημασία μέρα αυτή όσον αφορά την συνεργασία μας σε θέματα ασφάλειας. Συγχαρητήρια λοιπόν και σε όσους από εμά έχουν δουλέψει για αυτό το θέμα όλα αυτά τα χρόνια. 20 Νοεμβρίου είναι επόμενη συνεδρίαση στις 3 και στις 21 στις 9 το πρωί. Έληξη συνεδρίαση.